Καλώ welcome back ήρθατε λοιπόν. Περνάμε σημείο 8 τη ημερήσια ε, διάταξη το οποίο είναι προφανέ ε, ποιο είναι. Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ. Η τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ήταν στι 24 Μαΐου και η επόμενη θα είναι τον Μάρτιο του επόμενου έτου. Δεν ξέρουμε ακόμα την ημερομηνία. Οπότε καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Ο χρόνος βεβαίω μας πιέζει όλους. Βεβαίως... Ε, συνάδελφοι, δεν μπορώ να γράφω ενώ μιλάω στον κύριο Επίτροπο. multitasking capable? Μα δεν μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα μαζί. Ευχαριστώ και κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μεταξύ ημών για να ασχοληθούμε με ακρίβεια θα έλεγα σχετικά με την ατζέντα μας ως προς τις ε, χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι τα θέματα είναι σοβαρά. Οι οικονομικές αβεβαιότητες και αυτές είναι βαριές και παρατηρούμε διάφορα επεισόδια τα οποία εξελίσσονται από το 2008 και εντεύθεν. Αντιμετωπίζουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα, ενώ οι συνέπειες και τα ίχνη της κρίσης του 2008 ε, δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί. Και βεβαίως εξάγουμε συμπεράσματα από την κρίση αυτή και δεν πρέπει να έχουμε βραχία μνήμη λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές, οικονομικές, ε, πολιτικές συνέπειες, ε, την υπερχρέωση των κρατών, τόσο εδώ στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν σοβαρές προκλήσεις ταυτόχρονα και ασφαλώς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να είμαστε αποφασισμένοι και να κάνουμε αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο αποφασίζεται και σε επίπεδο των G20, αλλά και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 26 Οκτωβρίου. Και πρέπει λοιπόν να πράξουμε αυτό το οποίο αποφασίσαμε και να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα, αλλά και τον υπερβολικό παραλογισμό που υπάρχει όσον αφορά την αξιολόγηση των ε, χρεών χωρών εντός της ζώνης ευρώ. Η πολιτική θα πρέπει να ανακτήσει τα δικαιώματά της, τη θέση της, η οποία πρέπει να είναι πρώτη θέση θα έλεγα. Και οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εδράζονται σε τρεις άξονες. Απόκριση στην υπάρχουσα κρίση, ε, απαραίτητη ρύθμιση, αλλά και για μένα εξίσου σημαντικό μέτρα τα οποία έχουν σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Η παγκόσμια ανταπόκριση στην κρίση και αναφέρομαι στις δηλώσεις Μπαρόζο η Κομισιόν δηλαδή έδωσε, έδειξε το δρόμο, ένα φιλοπορία αν θέλετε, στη διάσκεψη κορυφής 26 και 27 Οκτωβρίου. Ήταν δύσκολο οι επικεφαλής, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να λάβουν αποφάσεις για όλες τις προκλήσεις. Το μέλλον της Ελλάδας, η διατηρησιμότητα του χρέους, η πρόκληση της υπερχρέωσης, η υποστήριξη των τραπεζών, η τήρηση των κοινών κανόνων, η διακυβέρνηση της ε, Ευρωζώνης. Το κάθε ένα από αυτά τα θέματα είναι τμήματα του μεγαλύτερου προβλήματος, ούτως ώστε να, ε, ε, να ξαναβρούμε το δρόμο της ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα μέτρα ε, βεβαίως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, να ληφθούν και να επιληθούν ε, εν μια νυχτή. Απαιτείται προσπάθεια από όλους, από τους ηγέτες. Ο φίλος και συνάδελφος Μάριο Μόντι βρίσκεται στις Βρυξέλλες ε, σήμερα και καλείται και αυτός να επιδείξει την αποφασιστικότητα που απαιτείται. Και με βάση όλα αυτά έρχομαι στο θέμα της ενίσχυσης των τραπεζών. Προτείναμε να ενισχύσουμε συστηματικά τις τράπεζες με ένα στρώμα υποστήριξης και προστασίας έκτακτο, πολύ υψηλού επίπεδου, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεσή τους στην ε, υπερχρέωση. Στο τελευταίο κοφίν σημειώσαμε πρόοδο ασχολούμενοι με λεπτομέρειες είναι σημαντικό και ξέρω ότι η Πρόεδρος ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για το θέμα της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ώστε οι τράπεζες να διαδραματίσουν τον πρωταρχικό ρόλο που είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το diverging, αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό εις βάρος της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Κάτι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζες ε, θα, θα πρέπει να διατηρήσουν την δυνατότητά τους ε, να ενισχύουν την οικονομία αλλά ε, αυτό το σχέδιο με τη βοήθεια των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί με βάση τις προτάσεις, τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προχωρήσουν στην επανακεφαλαιοποίηση με τον τρόπο τον οποίο περιέγραψα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την δυσκολία αυτή τη στιγμή της χρηματοδότησης των τραπεζών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και ε, γνωρίζουμε τις τα έκτακτα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για όλα αυτά. Αυτά είναι τα επίγοντα και όσον αφορά το σχέδιο έκτακτης αντίδρασης έτσι όπως αποφασίστηκε στις 26-27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν θέλουμε να ξαναβρούμε τη σταθερότητα, και να εξέλθουμε από την κρίση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τα διδάγματα του 2008 για μια πιο υγιή και πιο στέρεη βάση που απαιτείται για τον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω ρυθμίσεων. Είναι όρος εκ των ουκ άνευ αυτός για να εξέλθουμε από την κρίση. Αυτός ο κλάδος, ο χρηματοοικονομικός, είναι πολύ σημαντικός για μας. Άρα λοιπόν, περισσότερο παραποτέ έχουμε τη φιλοδοξία αλλά και την πρόθεση να να αναλάβουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο των G20, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του έτους η Κομισιόν θα ολοκληρώσει το έργο της των προτάσεων που θα θέσει επιτάπητος, δηλαδή το σύνολο των κειμένων που αναμένονται από πλευράς Κομισιόν ώστε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των G20 έχει διανεμηθεί ο πίνακας αυτών των προτάσεων. Σημειώνουμε πρόοδο, ταχεία και επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθώ στο κείμενο το οποίο βρίσκεται στη φάση της ε, τελικής ε, ολοκλήρωσης. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες ε, κείμενο το οποίο περιλαμβάνει πολλά αλλά πάνω απ' όλα την εποπτεία, την επιτήρηση. Και η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Κάθε εβδομάδα που περνάει βλέπω την ε, πρόοδο που σημειώνεται από όλες τις πλευρές. Απαιτείτε εσείς από πλευράς των Ευρωπαϊκών Αρχών έργο και χαιρετίζετε κάθε φορά την επίτευξη σύνθετων αποφάσεων. Το θέμα των, ε, της επίλυσης των swaps ε, είναι ε, ένα κείμενο στο οποίο καταλήξαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια των ασφαλίστρων κινδύνων. καταλήξαμε με μεγάλη προσπάθεια με τα ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα όσον αφορά στα παράγωγα. Ήδη η Κομισιόν της 14 Σεπτεμβρίου του 2010 υπέβαλε ε, τις προτάσεις της επί του short selling και εάν ε, υπάρξει συμφωνία με την παρέμβαση του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να είμαστε να, να προχωρήσουμε αρκετά και σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγγύηση των καταθέσεων. Ο Πίτερ Σάιμον καταβάλει προσπάθεια και πρέπει να προοδεύσουμε και οι Ευρωπαίοι αναμένουν πραγματική προστασία από μέρους μας. Γνωρίζω βέβαια τη δυσκολία του έργου του Ολσμιτ για την διασφάλιση ε, των ε, επενδύσεων και απαιτείται προσπάθεια και από δική μας πλευράς. Αυτά πολύ επιγραμματικά όσον αφορά το κείμενο. Ε, βεβαίως δεν λειτουργούμε μόνοι, υπάρχει, απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου. Επίσης, απαιτείται σειρά μεταρρυθμίσεων όπως είναι η τρίτη φάση της, της Βασιλείας. Η ε, πρώτη ζώνη του κόσμου μεταξύ των, υπογραφών ε, των υπογραφώντων την απόφαση του G20 είμαστε εμείς. Έχουμε την έκθεση Dot Marcaras και υπενθυμίζω ότι αυτό θα εφαρμοστεί σε 8.000 ε, τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια και λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης, ε, διότι στην Ευρώπη έχουμε ε, ομίλους τραπεζών. Και ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, ότι με την πρόταση αυτή παραμένουμε πιστοί στο πνεύμα και το γράμμα της Βασιλείας. Δηλαδή, επιτρέπουμε στους εθνικούς επόπτες να έχουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προχωρήσουν ε, πέραν της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο στην ατζέντα μας, την εβδομάδα που έρχεται. Πρόκειται για την αναθεώρηση της MIFID που εξυγχρονίζει τους όρους της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών. Ήδη συνεργαζόμαστε με τον Μάρκους Φέμπερ για την ολοκλήρωση αυτού του κειμένου. Το αναθεωρημένο κείμενο ως προς τις καταχρήσεις της αγοράς. Συνεργαζόμαστε με τον Αλέν Μακαρτή ως προς τα θέματα αυτά. Πέμπτο, πακέτο υπεύθυνων επιχειρήσεων. Οδηγία διαφάνειας με ιδιαίτερο τόνο και έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, την περασμένη εβδομάδα το Κολέγιο των Επιτρόπων υιοθέτησε ε, μία πρόταση σχετικά με τις οίκους αξιολόγησης. Ε, γνωρίζετε το προηγούμενο κείμενο, ο κύριος Κλίνς που ε, συνέταξε μία σημαντική έκθεση για να καταλήξουμε από αυτού. επί του θέματος αυτού δεν έχω καμία ιδεολογία, δεν είμαι υπέρμαχος καμίας ιδεολογίας. Δεν θέλουμε να βάλουμε εναντίον κανονός. Πρέπει να μετρούμε τον κίνδυνο των επιχειρήσεων, των ε, ιδρυμάτων, των κρατών. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ακρίβεια, αξιοπιστία και διαφάνεια, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα περασμένα χρόνια, διότι έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Ταυτόχρονα, οι αξιολογήσεις αυτές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία σας, δεν θα ε, πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουν εν κινδύνο την ε, σταθερότητα, ούτε και να δημιουργούν την εικόνα μιας υπερβολικής σταθερότητας. Δηλαδή αυτό αφορά τόσο τη μεθοδολογία, όσο και την διαφάνεια. Το, το μέγεθος των ευρωπαϊκών αρχών. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι η σύγκρουση ε, συμφερόντων, όπου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, με μια στενή προσέγγιση του 10% ας πούμε του κεφαλαίου κάθε ε, φορέα. Και εκεί θα πρέπει να διαφυλάσσεται η αστική ευθύνη αυτών των φορέων. Δουλέψαμε για να προχωρήσουμε και υπενθυμίζω ότι γνωρίζω τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι κανείς επίτροπος και βρίσκεται ενώπιον μιας ομάδας. Πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στην ομάδα μπορεί να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και θα πρέπει να αναζητηθεί μια μέση οδός. δού λοιπόν για κάποιες αποφάσεις χρειάστηκε να μας χρειάζεται περισσότερο χρόνος. Αλλά όσον αφορά λοιπόν τις, ε, τους οίκους αξιολόγησης, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στην ΕΣΜΑ, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών ε, Αξιών και αυτό θα πρέπει να γίνει με απόλυτα αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, διότι είναι και μία από τις βασικές μου φιλοδοξίες. Είναι η πρόληψη και η επίλυση της κρίσης των ε, τραπεζών, της τραπεζικής κρίσης. Ε, στόχος είναι η διάσωση τραπεζών που βρίσκονται σε κίνδυνο και όχι ε, να θέσουμε σε κίνδυνο τους ε, ε, φορολογουμένους. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάποιες αρχές που θα ισχύουν για όλες τις τράπεζες, αλλά θα υπάρχει ένας τρόπος στάθμισης για να μετρηθεί ο κίνδυνος, αν θέλετε, που διατρέχουν τα ιδρύματα αυτά. Και δεν θα πρέπει να σφάλουμε ως προς την κατάλληλη στιγμή αυτής της μεταρρύθμισης. Χρειάζεται να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ φιλοδοξιών και ρεαλισμού, ούτω ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτό το νέο καθεστώς το ταχύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι η πρόληψη σαφώς κοστίζει πολύ λιγότερο από την αποκατάσταση και θα έπρεπε και στην περίπτωση των τραπεζών να ισχύει αυτό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο συμβαίνει ε, αυτή τη στιγμή και αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά μια άλλη επιτροπή, τη νομική, αλλά θα υπάρξει μια πρόταση σε έναν άλλο τομέα που σαφώς θεωρείται ένα από τα θέματα υπομεταρρύθμιση είναι ο τομέας του ελέγχου, όπου και εκεί υπάρχουν και αποκλήσεις και εκεί απαιτείται διαφάνεια ώστε να αποκατασταθεί η ε, πίστη και η αξιοπιστία. Και θα βασιστεί στην έκθεση του κυρίου Ντεζάλγκο της 13ης Σεπτεμβρίου. Αυτά κυρίες και κύριοι πολύ συνοπτικά είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για θέματα, για ένα, μια ατζέντα πάρα πολύ ε, φορτωμένη με πολύ περιερχόμενο και με τη δική σας συμβολή και προσπάθεια θα επιτευχθεί. Ακούω πολλές φορές ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεραντέδρασε έναντι της ε, κρίσης. Το 2010 θεωρήσαμε ότι κάπως απομακρυνθήκαμε από την κρίση, από την κρίση αυτή των τραπεζών και των και ε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάπως χαλαρώσαμε και ξαναγυρίσαμε πίσω στο business as usual. Ωστόσο, ε, ήταν λάθος αυτό, διότι δεν πρέπει να έχουμε σύνδο, σύντομη, ε, ε, ισχνή μνήμη. Τώρα η κατάσταση επιδεινώθηκε και χρειάζεται πραγματικά αποφασιστικότητα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της ατζέντας. Η αποφασιστικότητά μου παραμένει άτρωτοι. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο των G20 για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην Ευρώπη με σειρά μέτρων που συνολικά πηγαίνουν πολύ μακριά και που έχουν το δικό τους ειδικό βάρος οφείλουμε και πρέπει να οικοδομήσουμε μια στέρεη βάση για το χρηματοοικονομικό οικοδόμημα και για την αγορά που έχουμε ανάγκη στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας. Πέραν των προτάσεων και θα τελειώσω σε λίγο, ε, αναφερόμενο στο πρόγραμμα του 2012, δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στους πολίτες, τους πολίτες καταναλωτές ή χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πιο κοντά στους πολίτες θα έλεγα με βάση το σύνολο των θεμάτων που προανέφερα. Με την πρωτοβουλία PRIPS θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών στις σχέσεις τους με τις τράπεζες και με τους άλλους ε, φορείς ε, 11 δις ευρώ καλύπτουν το σύνολο των επενδύσεων, τα διαρθρωμένα προϊόντα, τραπεζικά προϊόντα κλπ. Νομίζω ότι κάθε Ευρωπαίος επενδυτής θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος από τους ειδικού, ενημερωμένος ορθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα να καταλήξει σε αποφάσεις. εμπιστευόμενος τις αγορές. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα στις αρχές του 12. Δρομολογήσαμε την οδηγία τη MIFID, όπως επίσης και την οδηγία για την διαμεσολάβηση στις ασφαλίσεις. Όσον αφορά τους επενδυτές, πρότεινα ένα κάθετο κείμενο το οποίο αφορά στην τυποποιημένη πληροφόρηση των επενδυτών. Την προσεχή εβδομάδα θα κάνουμε μία πρόταση σχετικά με τα επενδυτικά κεφάλαια για να ενθαρρύνουμε τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ένας άλλος τομέας που θεωρώ ε, ότι είναι πολύ σημαντικός είναι αυτός του shadow banking υπήρξε μια έκθεση στους G20 της Κάνας. Βρισκόμαστε σε προκαταρτική φάση της χαρτογράφησης των πρακτικών και των νόμων που ισχύουν στην Ευρώπη. Μέσα στο 12 θα προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα και θα υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις. Πέραν των αποφάσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια στην αγορά αλλά και στον τραπεζικό τομέα. Αυτά κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, τα συμπεράσματα. Η βασική ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του χρόνου των αγορών, του χρόνου που τρέχει στις αγορές και της δημοκρατίας. Υπάρχει αστάθεια, υπάρχει έλλειψη σταθερότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχουν δομές οι οποίες εξασθένησαν εξαιτίας των υπερβολών του παρελθόντος και υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης. Έτσι λοιπόν απαιτείται έναντι των πολιτών που εσείς εκπροσωπείτε αποφασιστικότητα, αποφάσεις, ανακοινώσεις οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από ενέργειες, από πράξεις. Πρέπει να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία αποφασίζουμε. Πρέπει να εξηγήσουμε, και αυτό απαιτεί χρόνο, ότι το κείμενο που με μεγάλη προσοχή παρουσιάσαμε στην Κομισιόν στις 13-14 Σεπτεμβρίου του 2010 πρέπει να εξηγήσουμε ότι ε, ε, αυτό συμβαίνει 12, 13, 14 μήνες μετά. Αυτό οφείλεται στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πάντως έχω την εντύπωση ότι όταν εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελέσματα, δίνουν καρπούς και αυτό είναι προφανές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χωρίς τη δική σας ε, υποστήριξη βεβαίως δεν πρόκειται να πετύχουμε και να καλύψουμε αυτή την ατζέντα και να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να αποκατασταθεί δηλαδή αυτή η χρηματοοικονομική σταθερότητα που είναι απόλυτη ανάγκη για να υπάρξει βάση για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, του ανταγωνισμού και της ε, ε ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν πολλά θέματα για τις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες. Πολλοί είναι οι ομιλητές και αν θα σας αναφέρω να μου το πείτε. Ο Ζαν Πολ κάτι θέλει να πει. Αρλίν. Yes, uh, Vicky, you και εσύ θέλεις να μιλήσεις, Βίκη, γιατί η Κέι δεν είναι εδώ. Ο Φιλίπ, γιατί ο Σβέν δεν είναι εδώ. Ο κύριος Χουντής. Okay, Pascal first. Πρώτα Πασκάλ. Then, um, Μετά. Ο κύριος Χουντής. Μετά Φιλίπ. Μετά Λίαν. Μετά ο Διόγκο, Λεωνάρτο και η Ελίσα. Υπάρχει κάποιος άλλος τον οποίο δεν ανέφερα. Ωραία, πλήρης ο κατάλογος. Ο Ζαν Πολ Γκοζές έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θα σας υποβάλω ερωτήσεις. Σας το λέω εξ αρχής, γιατί ίσως θεωρηθεί ότι συμφωνήσαμε εκ των προτέρων. Και η απάντηση θα πλεόναζε. Δεν έχουμε όλη την ίδια εντύπωση, λέει ένας ομιλητής. Εν πάση περιπτώσει, ως προς την εισήγησή σας, ε, μιλήσατε για αυτή τη γενική ιδέα. Λέμε ότι ο χρόνος της δημοκρατίας δεν συμπίπτει με τον χρηματοπιστωτικό χρόνο, όμως ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να διευθετήσουμε και τα περί και τα περί χρηματοπιστωτικών. Όμως οι πολιτικές αρχές, ε, εάν δεν εποπτεύσουν σωστά, δεν θα καταφέρουμε τίποτα ενώπιον τον Μπαρόζο και Βάνο Ρομπό είπα στην Ολομέλεια ότι οι αγορές ποτέ δεν θα ικανοποιηθούν διότι από τη φύση τους ε, απεχθάνονται τον κίνδυνο και την έλλειψη ασφάλειας γιατί διαφορετικά η ανασφάλεια και ο κίνδυνος ε, μεταβιβάζονται. Θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει κάθε μέρα προβάλλει κάθε μέρα νέες ιδέες, ευρωμόλογα, γίνεται λόγος για αυτά, η Σιλβή θα επανέρθει. Γιατί όμως η Κομισιόν δεν προχωρά μέχρι τέλους στη σκέψη της. Μιλάμε για οίκους πιστοληπτικής ικανότητας και μπορώ να σας πω ότι προσωπικά και με την υποστήριξη του ΕΛΚ και πολλών άλλων θα υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της σκέψης της Κομισιόν. Έχει σημασία και η σκέψη αλλά και η δράση πρωτίστως. θα πρέπει να βρούμε ένα καθεστώς για τις χώρες της Ευρωζώνης που γνωρίζουν μεγάλες δυσκολίες και σαν να βρισκόμασταν σε μια ομοσπονδία θα πρέπει να βρούμε ρήτρες προστασίας γιατί δεν ζούμε σε μια ομοσπονδία. Θα μιλούσαμε για ένα κεφάλαιο 11 της Ευρωζώνης αν μιλήσουμε υπό αγγλοσαξονικούς όρους. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι θα πρέπει να αναστείλουμε τη βαθμολόγηση, αλλά δεν θα πρέπει να δίνουμε σημασία στις φημολογίες. Όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης, γνωρίζετε πολύ καλύτερο από μένα πόσες προσπάθειες έπρεπε να καταβάλουμε, έτσι ώστε η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, να μπορεί να δράσει έναντι των οίκων και μπορώ να πω δημοσία ότι ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ ήρθε να με βρει στις 18 Οκτωβρίου και δεν μου είπε πότε θα συμφωνούσαν οι τρεις οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας και αυτό έγινε στις 31 Οκτωβρίου και οι εθνικοί ρυθμιστές ε, αναλαμβάνουν δραστηριότητα. Σήμερα οι οίκοι αξιολόγησης πρέπει να τύχουν εποπτείας. Ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ είπε ότι ίσως θα έπρεπε να μειωθεί αυτή η εποπτεία, όμως το είπα ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών σας υποστηρίζει. Πιστεύει ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια ευφυή ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν ρυθμίζουμε για να ρυθμίσουμε. Το χρειάζεται η οικονομία. Θα πρέπει να ορίσουμε και να περιορίσουμε περισσότερο τους κινδύνους για το καλό της οικονομίας. Ο Επίτροπος θα απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πως εγώ θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τις ε, επιθέσεις που δέχεστε από τον ε, Βρετανικό τύπο. Να σας αναφέρω μόνο έναν τίτλο, ο Μπαρνιέ εναντίον ε, των Βρετανών. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι αντίπαλός σας, αλλά εταίρος για να δημιουργήσουμε ένα πιο ανοιχτό και διάφανο οικονομικό σύστημα στην Ευρώπη. Τούτου λεχθέντος βεβαίως θα πρέπει να τονίσω πως καλωσορίζει το έργο σας που κάνετε στην τρίτη οδηγία κεφαλαιακής επάρκειας και την εφαρμογή της και καλό είναι το ότι ε, αφιερώνετε το χρόνο σας για να δείτε τα... θα μας βοηθήσετε να δείτε τα της εφαρμογής. Η ερώτησή μου είναι τι σκοπεύετε να κάνετε με τα κρατημέλη που δεν εφαρμόζουν την τρίτη οδηγία κεφαλαϊκής επάρκεια. Επίσης να τονίσουμε στις τράπεζες τη στιγμή που ετοιμάζονται να δώσουν τον πόνους πως ε, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσει αυτής της ε, οδηγίας και βεβαίως να προτιμήσουν τη ρευστότητα από τις ε, αμοιβέ και είναι σαφής η οδηγία σε αυτό. Και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας το ότι σήμερα μάλιστα ε, η Επιτροπή Υψηλών Αμοιβών στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε την έκθεσή της και τις συστάσεις της όσον αφορά τη διαφάνεια και την ε, εταιρική διοίκηση και να πω σε κάποιους στην Επιτροπή το ότι δεν γνώριζα πόσο επικεφαλής της ε, Barclays τα τελευταία 20 χρόνια πήρε μια αύξηση 5.000% στην Λόιτζη, η οποία πλέον ανήκει στο κράτος, μιλάμε για την ίδια 20 ετία, μια αύξηση 3.000% και γενικά βεβαίως οι κορυφαίοι στις ε, τράπεζες ε, πληρώνονται από 70 μέχρι 500 φορές περισσότερο από τους απλούς ε, εργαζόμενους. Ε, πρέπει να το δούμε αυτό και να αντιληφθούμε πως πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από προγράμματα λιτότητας, χάνουν τις δουλειές τους και δεν είναι αυτό το σωστό μήνυμα σε καιρούς ε, λιτότητας όταν κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν μυαλά. Και να πω πως εκτιμώ το έργο που κάνετε στον τομέα αυτόν. Σιλβί. Η Σιλβί. Ευχαριστώ Επίτροπε, σας ευχαριστώ γιατί βρίσκεστε εδώ για να συνεχίσω σε αυτά που είπε ο Ζαν Πόλος προς τα ευρωομόλογα. Μην λέτε ότι παίρνουμε πολλές πρωτοβουλίες. Θα σας υποστηρίξουμε όταν ε, προωθείτε αυτή τη συλλογιστική. Δηλαδή δεν σπέβδουμε να φτάνουμε σε συμπεράσματα, φτάσουμε σε συμπεράσματα ως προς αυτό το σκέλος. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σκιαγράφηση για να δούμε τι έχουμε ενώπιόν μας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εσάς και την Επιτροπή. Όχι ως προς το νομοθετικό σκέλος, αλλά ως προς τη συνεχή αξιολόγηση. Από την εποπτεία αναρωτιόμαστε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά ως προς την οικονομική διακυβέρνηση θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα κείμενα, λέμε δηλαδή ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες για το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά ε, συμφωνούμε επί του περιεχομένου. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως δεν θα πρέπει να επαγρυπνούμε ως προς την εφαρμογή, πέρα από τις αλλαγές, δηλαδή να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι αποφάσεις μας, το νέο βαθμολόγιο, τι θα γίνει με αυτό, με την πειθαρχία που υπάρχει ως προς τον τραπεζικό έλεγχο, την εκ νέου κεφαλαιοποίηση, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα πιο δημιουργικό θεσμικό παιχνίδι έτσι ώστε πέρα από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο οι πολίτες να νιώθουν ότι πραγματικά γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το τι μέλη γενέστε. Έχετε μια φορτωμένη ατζέντα γιατί καθυστερήσαμε εδώ και πολύ χρόνο, χρόνο. Άρα κατανοούμε το ότι υπάρχει υπερρύθμιση, αλλά ίσως χρειάζεται ένα πιο μακροχρόνιο εγχείρημα επαλήθευσης και εποπτείας της εφαρμογής των κανόνων. Ο τρόπος θα απαντήσει στις τρεις αυτές ερωτήσεις. Νομίζω και θα ήθελα να πω προς τον Ζαν Πολ Γκοζές αλλά και προς τον καθέναν αν και δεν ήθιστε, οι χρηματοοικονομικές αγορές θα πρέπει να δεχτούν τη δημόσια ρύθμιση. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Θα πρέπει να γίνει αυτή η δημόσια ρύθμιση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η οποία δυστυχώς αποτελούσε μεγάλο έλλειμμα μέχρι τούδε. Ως προς τους χρηματοοικονομικούς φορείς έχουν δίκιο όταν ζητάνε μία σταθερότητα, γιατί όποια επιχείρηση κι αν έχουμε πρέπει να έχουμε σταθερούς κανόνες. Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό θα πρέπει να τα κάνουμε όλα παράλληλα και να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Κατανοώ αυτά που είπε ο Ζαν Πολ Γκοζές για τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Διαβάζω κι εγώ τον τύπο και θα ήθελα να πω στην άλλη Μακάρτη ότι διαβάζω και τον Βρετανικό τύπο. Θα ήθελα να σταθούμε στην κοινή μας εργασία επί της ουσίας. Πέρα από αυτά που ελέγχθησαν, επιπροσθέτως είχα προτείνει κάτι το συγκεκριμένο, όπως είχε πει και το Δούνο του, δηλαδή ε, να γίνεται αναστολή βαθμολόγησης μέχρι ότου και η ΕΣΜΑ αποφανθεί για ορισμένες χώρες οι οποίες την χάνουν ευρωπαϊκής υποστήριξης και διεθνούς υποστήριξης για να μην προσθέσουμε στην αστάθεια που ήδη υπάρχει. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και ίσως θα πρέπει αυτό να το εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όπως είπε ο Ζαν Γκοζές. Ως προς ανοιχτές πωλήσει, δεν είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφαίνεται ή ολοκληρώνει τις προτάσεις της Κομισιόν. Σήμερα η ΕΣΜΑ εποπτεύει 30 οίκους που έχουν ε, ενταχθεί και εγγραφεί και ορίζουμε το γενικό πλαίσιο κανόνων. Θα ήθελα να πω προς τον ότι υπάρχουν και διαφοροποιημένες θέσεις. Εγώ υποστηρίζω τον κύριο Μάγιορ και τους άλλους υπευθύνους οι οποίοι με περιορισμένα μέσα προσπαθούν κάτι να κάνουν. Αυτό αφορά και τις είπα. Είδατε τι έγινε στο Κογκρέσο ως προς τη συζήτηση για τη μείωση του ρόλου των εποπτικών αρχών. Και αν οι ανεξάρτητες ε, αρχές δεν μπορούν να λειτουργήσουν, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να δουλέψει κανείς. Εμείς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΜΑ και με τις άλλες αρχές κινητών αξιών και επιβεβαιώνω την εμπιστοσύνη μου προς αυτές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας ως προς την ανάληψη πρωτοβουλειών. πριν από τη Standard Poor's στη βαθμολόγηση ως προς ένα κράτος μέλος, δεν το είχαμε λάβει υπόψη σοβαρά. Τότε διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι οίκοι είχαν συνδρομητές επιπληρωμή που λάβαναν πληροφορίες πριν από τους άλλους. Αυτό είναι λογικό. Δηλαδή να υπάρχει προτιμησιακή σχέση με ορισμένους πελάτες, με μια συγκεκριμένη πελατεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επιτείνει και τους κλειδονισμούς της αγοράς. Αυτό θα το δούμε και στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας και ευχαριστώ τον Ζαν Πολ για τα εθνικά του λόγια. Η κυρία Μακάρτη μίλησε και στάθηκε σε ορισμένες επικρίσεις που δέχομαι. Έχω πρόβλημα με τους Βρετανούς και όχι μόνο στον τύπο. Ένας ε, Γάλλος, λένε, διορίστηκε επίτροπος της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα πρέπει να σας αποθαρρύνει το γεγονός ότι ένας Γάλλος ορίστηκε, ορίστηκε, διορίστηκε επίτροπος εσωτερικής αγοράς, αλλά αυτό που θα έπρεπε να σας εκπλήξει είναι ότι εδώ και 60 χρόνια δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Στο. Ο ρόλος του City είναι πολύ σημαντικός. Είναι μεγάλη τύχη για την Ευρώπη ότι με το Λονδίνο έχουμε αυτή τη συνεργασία. Και το City έχει προσαρτηθεί στην Ευρώπη στην Ήπειρο δηλαδή, παρά αλλού. Έρχομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα με το ΣΥΤΙ για να ολοκληρώσουμε αυτή την ε, χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Δυστυχώς ε, και το ΣΥΤ ήταν ευάλωτο, κατέστη πιο ευάλωτο από την χρηματοοικονομική αυτή κρίση και θα πρέπει να έχουμε μια ε, δυνατή μια στεναρή βάση και γι' αυτό ακριβώς σε όλα τα κείμενα που εγκρίναμε η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ε, είχε συμφωνήσει καθ' ολοκλήριαν. Ως προς το CRD, για την οδηγία για τις ε, κεφαλαιακές απαιτήσεις τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί διαδικασία επί κατά αρκετών κρατών τα οποία ακόμα δεν, μας, ε, δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία αυτή στο εθνικό δίκαιο. Δεν έχει ενταχθεί στην εσωτερική ένωμη τάξη τους. Ως προς το θέμα της κυρίας Μακάρτη για τις... Ε, για στο CRD, θα ήθελα να πω ότι η οδηγία 3 για τις κεφαλιακές απαιτήσεις θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να δούμε πώς καταβάλουν τα άσφα, πώς έχουν οι αποδοχές, ποιο είναι το πλαίσιο αποδοχών και δεν νομίζω ότι αρκεί μόνο να μιλήσουμε για σύνεση έτσι ώστε να μην γίνουν καταχρήσεις. Και αυτό αφορά και τα μπόνους που δίνονται που δεν δικαιολογούνται ενώπιον του πολίτη και ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Εργάζομαι επ' αυτού, αλλά με απόλυτη σοβαρότητα θα πρέπει να προχωρήσουμε Περαιτέρω και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27ης Οκτωβρίου είπε να μην χορηγηθούν, να μην αποδοθούν μπόνους σε καμία από τις συστημικές τράπεζες. Και ιδίω μέσα στα πλαίσια αυτού του 9% που αναφέρθηκε. Η Σιλβι Γκουλάρ μίλησε για τη σωρία κειμένων που έχουμε, για την πληθώρα κειμένων αυτή η απόφαση ελήφθη σε επίπεδο G20, στο ανώτατο επίπεδο οικονομικής διακυβέρνησης. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για πλήθος εγγράφων. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για το κείμενο ως προς την εποπτεία γιατί έχω και την ατζέντα της εσωτερικής αγοράς, μην το ξεχνάτε αυτό. Ίσως χρειαστεί κρατούν ε, ορισμένες μέρες, δηλαδή μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, έτσι ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση και τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα, δηλαδή εύληπτα περισσότερο. Ως προς την αξιολόγηση, γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ε, διαδραματίσει ένα συγκεκριμένο ρόλο, διότι πέρα από τη σωρία ρυθμιστικών κειμένων, όπως είπε η κυρία Γκούλαρ, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το πακέτο των έξι νομοθετημάτων. Τι θα γίνει μέσα στη διαδικασία προϋπολογισμού, διότι θα προβάλλουμε λειτουργικές ε, προτάσεις για την δημοσιονομική εποπτεία. Χρειάζεται μία ε, δημοκρατική εποπτεία, ένας δημοκρατικός έλεγχος. Ξέρω τι λένε για τους επιτρόπους, τι λέγεται για τους επιτρόπους. Πολλές φορές γίνεται λόγος για μία τεχνοκρατία, αλλά εμείς έχουμε νομιμότητα, ιδιαίτερα ενώπιον σας. Μιλάμε για δημοσιονομικό έλεγχο στα κράτη ε, μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης, της κοινή διαχείρισης του ευρώ. Χρειάζεται λοιπόν δημοκρατικός έλεγχος σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων όπως και του ευρωπαϊκού. Εν πάση περιπτώσει, η σωστή εφαρμογή και η αξιολόγηση, πώς θα γίνει, θα το σκεφτώ, κυρία Γκουλάρ, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εξεύρουμε ένα συλλογικό πλαίσιο ελέγχου. Επειδή πιστεύω ότι αυτή η ατζέντα ρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρωθεί, θα χρειαστούμε ένα χρόνο ακόμα. Το δεύτερο τμήμα της εντολής μου, πέρα από ορισμένα κείμενα υπέρ του καταναλωτή θα αφορά την επικαιροποίηση κειμένων και τη σωστή εφαρμογή όλων αυτών των κειμένων. Αυτά μπορώ να σας πω. για την σωστή εφαρμογή και αξιολόγηση των κειμένων. Μιλάμε και για νέα μέσα για ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια καλή αξιολόγηση των κειμένων και μια σωστή ρύθμιση. Ευχαριστώ. Πράγματι μου φαίνεται πως ε, η εφαρμογή, η επιβολή πρέπει να γίνει τόσο ενδιαφέρουσα όσο η νέα νομοθεσία. Και πρέπει νομίζω και η Κομισιόν να ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το ζήτημα όσο ασχολείται με την νέα νομοθεσία και χαίρομαι που επιμένουν σε αυτό οι συνάδελφοι. Κατόπιν, Πασκάλ Καμφέν, ε, κύριο Χουντή και Φιλίπ Λαμπέρτ. Πασκάλ. Και, και η Βίκη, να ακούσουμε τέσσερι. Ωραία, η Βίκη πρώτη. Ευχαριστώ, Σάρων. Μιλάμε για την ανάπτυξη πολύ και πρέπει να το εννοούμε γιατί είμαστε σε καιρούς ε, πολύ χαμηλής εμπιστοσύνης ε, και στις αγορές και ε, στους καταναλωτές. Κάποιες ερωτήσεις για την οδηγία ξέρετε πως ή βάλαμε κάποια διατύπωση για να εξαιρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο. Δεν ξέρω εάν ε, αυτό ισχύει και θα ήθελα να μας ε, βοηθήσετε για τα στεγαστικά δάνεια. Εάν ακούσουμε όλες τις προτάσεις εδώ πέρα, κινδυνεύουμε όλο, όλα τα στεγαστικά δάνεια σε ολόκληρη την Ευρώπη να απαιτεί να έχει όλες τις πιθανές επιλογές σε οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό μάλλον ακριβό μου ακούγεται. Ναι, συμφωνώ μαζί σας να σταματήσει ο ανεύθυνος δανεισμός, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, αλλά να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε και το κόστος. Αλλιώς δεν θα έχουμε ανάπτυξη καθόλου για το θέμα του σύφης που αναφέρατε μόνο αυτοί θα έχουν πρόσβαση στις ε, κεφάλαια αγορές και βεβαίως ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος και μετά για το θέμα της οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων. Συμφωνώ πλήρως πως χρειάζεται χρειάζονται οι ίδιοι κανόνες. Συμφωνώ πλήρως πως ο ορισμός του κεφαλαίου των ε, στοιχείων ενεργητικού και της στάθμισής τους πράγματι πρέπει να έχουν διαφάνεια. Δεν συμφωνώ πως κάθε χώρα πρέπει να έχει όμως το ίδιο επίπεδο του λόγου αυτού και Συμπτωματικά μαζί μου συμφωνεί ο Μάριο Ντράγκη, ο κύριος Τρισέ όταν ήταν διοικητής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, διάφορα κράτη-μέλη και ο κύριος Ντελαροζιέ στην ε, αρχική του έκθεση. Οπότε κύριε Επίτροπε ξαναδείτε μαζί μας πού χρειάζεται να έχουμε ενιαίους αγώνες, α, κανόνες γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για χώρες εντός της Ευρωζώνης, ειδικά για χώρες οι οποίες δεν μπορούν να ελέγξουν το επιτόκιό τους, να μπορούν να χρησιμοποιούν μακροπροληπτικά μέτρα κατά των διαφόρων φουσκών αυτών. Σας ευχαριστώ, Πασκάλ. Τρία σχόλια και ερωτήσεις, πολύ γρήγορα. Πρώτον, το Leveraging. Lever, μόχλευση. Απομόχλευση. Οι τράπεζες ε, έχουν βεβαίως ανάγκες σε ίδια κεφάλαια και αντί να αναζητήσουν ε, επιπλέον ίδια κεφάλαια, εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους. Και αυτό βεβαίως έχει τις συνέπειες του στην πραγματική οικονομία κλπ. την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου αποφασίστηκε να υπάρξει μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε οι τράπεζες να διασφαλίσουν αυτή την μείωση των ιδίων πόρων. Έκτοτε, καταρχήν το πράγμα επήγει ούτως ή άλλως και πιστεύω ότι η απόφαση αυτή, την απόφαση αυτή δεν την, η απόφαση αυτή δεν ακολουθήθηκε από την ίδια την πραγματικότητα. Ποια είναι λοιπόν η απόφαση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή και η Κομισιόν θα παίξει ρόλο σε αυτό το βασικό θέμα, ούτω ώστε η απομόχλευση, deleveraging, να ε, γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τρόπο κανονικό και όχι άτακτο. Δεύτερο σημείο, πολύ γρήγορα, αφορά τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου. Ευχαριστώ για τα σχόλια τα οποία κάνατε σχετικά με την ολοκλήρωση του φακέλου, σχετικά με τα ασφάλιστα κινδύνου και σας ευχαριστώ και για το ρόλο που διαδραματίσατε στην αναζήτηση μιας συμβαστικής λύσης. Το κείμενο βεβαίως ασχολείται με την αγορά των των κινδύνου, όχι με την έκδοση. Ένας όμως από τους κινδύνους ή από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι κανόνες πρόνοιας καλύπτουν το κίνδυνο με τα CDS, τα οποία όμως δεν έχουν εκδοθεί από φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν και τον ίδιο βαθμό κινδύνου. Και σε όλες τις πολιτικές ομάδες αυτό εντοπίστηκε ως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει απάντηση λοιπόν και ε, ακόμα και αν υπάρχουν επιτάπητος 29 κείμενα όπως ανέφερε η Πρόεδρος Ενδεχομένως λείπει ένα κείμενο όσον αφορά τις, ε, τους κανόνες αυτής τους ε, προληπτικής εποπτείας, αν θέλετε. Και είναι απολύτως απαραίτητο να λυθεί το πρόβλημα αυτό σήμερα, διότι πάρα πολύ γρήγορα αυτό θα συνδεθεί με τα ε, παράγωγα προϊόντα και θα έχει άλλες συνέπειες, είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε πάλι μαζί μας εδώ. Εκτιμώ τις προσωπικές σας προσπάθειες ε, που κάνετε και εκτιμώ ότι δίνετε και σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω σε αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και μία ερώτηση για να μου δώσετε κάτι απάντηση αν μπορείτε σήμερα. Το σχόλιο. Ενδιαφέρονται αυτά που μας είπατε. Σε μια στιγμή που η κρίση σοβεί υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωζώνη και όλα αυτά που γνωρίζουμε και βιώνουμε αυτές τις μέρες. Ακούω, άκουσα και από εσά μια δικαιολογία και από άλλους ε, κομισάριους ότι ο χρόνος των αγορών τρέχει πιο γρήγορα από το χρόνο της δημοκρατίας, της πολιτικής, των θεσμών. Επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι αυτή είναι μια πολύ εύκολη απάντηση, πολύ εύκολη απάντηση, δεν εξηγεί γιατί η Κομισιόν πάντα φτάνει καθυστερημένα και όταν φτάνει μάλλον προς λάθος κατεύθυνση δουλεύει. Το δικό μου σχόλιο είναι και μιλώ γενικά για την Κομισιόν, δεν μιλάω προσωπικά για σας, ή δεν μπορείτε ή δεν θέλετε ή και τα δύο. Δεσμευμένοι, θα σας εξηγήσω πώς το ερμηνεύω εγώ, από ιδεολειψίες και θεωρίες που μας οδήγησαν στην κρίση αλλά η συνταγή συνεχίζεται. Ένα παράδειγμα για να μην θεωρηθεί ότι έχω εύκολο αντιπολιτευτικό λόγο. Τι γίνεται με τους οίκους αξιολόγησης. Τώρα θυμηθήκαμε και ακόμα δειλά αυτά τα μέτρα όταν από το 2009, τουλάχιστον στο επίπεδο της Ευρωζώνης, εξέφρασαν την επιθετικότητά τους και την αναξιοπιστία τους με αρχή την Ελλάδα, όταν μετά το ξεδίπλωμα της κρίσης και την ευθύνη που είχαν καθώς οδηγούσαν τους επενδυτές στη Lehman Brothers, έσπευσε η Κομισιόν να διορθώσει ένα σωστό κανονισμό και να τους ξανακάνει νοικοκυρέως, να τους ξανακάνει επιδιαιτητές, να τους ξανακάνει εκτιμητές και μάλιστα των οικονομικών των χωρών. Και φτάσαμε αυτό που φτάσαμε και έχω στα αυτιά μου ακόμα την οργισμένη τελευταία δικιά σας κραυγή κατά των οίκων αξιολόγησης. Και το δεύτερο εισαγωγικό για μια ερώτηση και θα τελειώσω. Ξέρετε στη χώρα μου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λένε στην κρίση φτάσαμε εδώ, φτάσαμε εκεί, φτάσαμε εκεί. Έγιναν και σκάνδαλα και επιτέλους κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί κάπου πρέπει να υπάρξει μια αξιοπιστία. Έρχομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιά σας ως ε, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς. Δεν θα, ρωτήσω πάλι για τον ΟΤΕ, για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, θα σας ευθυνδιάσω. Θα μου δώσετε μια απάντηση γραπτή, τα είπαμε στην Ολομέλεια, δεν θέλω να τα ξαναλέμε αυτά. Θέλω να σας βάλω το γενικότερο ερώτημα και αυτό τελειώνει. Υπάρχει το πρόβλημα των δημοσίων συμβάσεων Υπάρχουν καταγγελίες ότι μεγάλες εταιρείες Siemens, Siemens MAN δωροδόκησαν κρατικούς αξιωματούχους για να πάρουν τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν έχω υπόψη μου, βοηθήστε με, αν έχει γίνει κάποια έρευνα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν έχετε βγάλει κάποια πορίσματα, αν έχετε κάποιο σχέδιο αποκατάστασης των κοινοτικών κανόνων, αν έχετε βγάλει κάποιο σχέδιο υπεράσπισης των χρημάτων της Ένωσης, γιατί πολλά από αυτά τα χρήματα είναι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες, επιτέλους κάποιοι πρέπει να πληρώσουν και σε αυτό το επίπεδο. Κυβερνήσεις πέφτουν, πρωθυπουργοί αλλάζουν, όλα αυτά. Σε αυτό το επίπεδο τι σκεφτόσαστε να κάνετε, τι ευθύνες υπάρχουν, πώς μπορεί να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, 17 ερωτήσεις, 4 σχόλια και δεν ξέρω πόσα σχόλια. Αλλά θα περιοριστώ σε ένα σχόλιο, σε μία ερώτηση. Είπατε ότι ο χρόνος της δημοκρατίας δεν είναι ταυτόσιμος με το χρόνο των αγορών. Ως προς το CRD, δηλαδή Οδηγία Κεφαλαιοκών Απαιτήσεων Επάρκειας 4, CRD 4, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Έχουμε το θέμα του ΣΥΦΙΣ και το CRD4 είναι ακριβώς το όχημα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συστημικά προβλήματα. Δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει κάτι το οποίο και για μια φορά θα συμφωνήσω με τους Βρετανούς, οι ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας προτείνουν να υπάρξει διαχωρισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Και νομίζω ότι είναι πια καιρός να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά επίσης και σε εμά. Σε εμά, όταν λέω βεβαίω η Βρετανία είναι σε εμά επίσης, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοώ στην ε, Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επειδή αναφερθήκατε και στο shadow banking, ε, διότι ένας τρόπος καταπολέμησης του shadow banking είναι ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε τις προβλέψεις της οδηγίας κεφαλαϊκών πετήσεων ε, κεφαλαϊκής επάρκειας, για να αποκαλύψουμε τις δραστηριότητες του shadow banking. Άρα λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όχημα του CRD4 και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και χρόνο ε, αντί να πολλαπλασιάζουμε τα νομοθετικά κείμενα. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας άποψη από αυτού και τις άλλες ερωτήσεις μου δεν θα τις υποβάλω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Με μία φράση θα συμπληρώσω την απάντηση που έδωσα στην Σιλβή. Υπάρχει ένα μέσο, ένα εργαλείο το οποίο θα μας είναι πολύ χρήσιμο στο έργο μας. Διότι ε, θα, υπάρχει, θα υπάρχουν σορευμένες επιπτώσεις και αποτελέσματα από την θέση σε ισχύ αυτών των κειμένων το προσεχές έτος και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και την επίδραση όλων αυτών. Ένα άλλο θέμα στο οποίο δουλέψαμε πολύ είναι και η επαλήθευση της ε, η επαλήθευση της στάθμισης των όσων κάνουμε με τους άλλους, δηλαδή την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αν πραγματικά βρισκόμαστε σε παράλληλο δρόμο, παράλληλη γραμμή ή όχι. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν σχετικά με την ανάπτυξη, ότι δηλαδή ένα βασικό σημείο κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Και βεβαίως εδώ είναι πολύ σημαντική αποφασιστικότητα που πρέπει να επιδείξουμε και δεν με εντυπωσιάζουν οι εκστρατείες lobbying παρά το γεγονός ότι τις παρακολουθώ. Και απαιτείται ρύθμιση το ταχύτερο δυνατό ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη. Ως προς το προοπτικές Και πάλι, ε, αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια, είναι τα πρότυπα. Θα δείτε ότι συστηματικά, χωρίς να τίθεται να αμφιβόλο ο βαθμός διαφάνειας που υπάρχει, όπως ακριβώς είχα δεσμευθεί ενώπιόν σας, θα ε, ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες τις σχετικές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε και μια διαβούλευση με τους υπευθύνους των χρηματιστηρίων της Ευρώπης, ούτως ώστε να υπάρξει μια διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να δούμε ποιο μοντέλο, ποιο πρότυπο θα είναι πιο χρήσιμο, είτε αυτό των σκανδιναβικών χωρών, είτε της Γερμανίας, είτε άλλων. Σχετικά τώρα με τα στεγαστικά. Ακόμα το κείμενο είναι υποσυζήτηση σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια. Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και από πλευράς Βρετανών. Δουλεύουμε λοιπόν με σκοπό να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο σταθερό και ευρωπαϊκό, το ταχύτερο δυνατό. Τώρα, ως προς το CRD4, όπου εκεί το επίπεδο ευελιξίας που απαιτούν κάποιες χώρες για να αντιμετωπίσουν ας πούμε συγκεκριμένες ε, δυσκολίες ή προκλήσεις ας πούμε στεγαστικά ή όμιλοι ε, τραπεζών κλπ. Και προβλέψαμε στο κείμενο της 20ης Ιουνίου τις ευελιξίες, τις ευελιξίες των λέει οι που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης, ε, αυτών των συγκεκριμένων προκλήσεων. Τώρα, το θέμα της ε, αγοράς των ακινήτων ποικίλει από χώρα σε χώρα και εκεί απαιτείται ε, μία εποπτεία για να καλυφθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν φορέας ή φορείς που βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή επικράτεια ενδεχομένως να απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια με την ε, χρησιμοποίηση αυτού που αποκαλούμε ένα στρώμα προστασίας. Από την άλλη, απαιτούνται κανόνες ε, προληπτικής εποπτείας, πολύ αυστηρότεροι τέτοιοι κανόνες, για να επιτευχθεί η σταθερότητα. Μέσα από αυτά τα μέσα χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοηδία, ή άλλες χώρες θα μπορούν να ε, εφαρμόσουν επιπρόσθετους μηχανισμούς εποπτείας αν αυτό το κρίνουν απαραίτητο. Αυτό είναι απολύτως δυνατό, αν η Βρετανική κυβέρνηση το αποφασίσει στο πλαίσιο των αποφάσεων CRD4. Να πω το εξής θέλουμε να δουλέψουμε στο πλαίσιο αυτών που, ζητή, που μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ενιαία αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι ένα ευρύτερο θέμα. Όχι, δεν μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ δεν μιλούσα για το Ηνωμένο Βασίλειο, διακόπτη κύρια. Όχι, και εγώ απάντησα ότι μίλησα και για άλλες χώρες, ας πούμε τη Σουηδία. Δεν έχω πρόβλημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χώρα εκείνη η οποία ε, εφλέγεται λέγοντας ότι αυτά τα οποία προτείνονται δεν είναι επαρκώς ευέλικτα. Το ίδιο ισχύει όμως και για την Σουηδία και μίλησα και με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας. Ίσως αυξηθεί ο βαθμός ευελιξίας. Αυτό όμως που θέλω είναι να ε, σεβαστούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν δεν πρόκειται να δεχθώ 27 διαφορετικά τραπεζικά συστήματα. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να αναπτύξω σε συνεργασία με εσάς μια ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν η κανονιστική αρχή στη Σουηδία αποφασίσει ότι θέλει επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση ας πούμε κινδύνων από τις χώρες της Βαλτικής θα είναι απολύτως ελεύθερη η αρχή αυτή να το πράξει. Δεν θα πω όμως σε λεπτομέρειες για τις δυνατότητες αυτές. Για το θέμα της απομόχλευσης. Βλέπουμε να επιταχύνονται τα πράγματα και πρόκειται για μια ανησυχία που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, την Παρασκευή είχα μια συνάντηση με τον κύριο Ενριάτ που είναι ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Φορέα. Θέσαμε και σε αυτόν το ερώτημα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων λοιπόν που του δώσαμε και που μπορεί να ενισχυθούν στο μέλλον, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των και των εθνικών εποπτικών αρχών υπάρχουν δεσμεύσεις και αυτές θα πρέπει να μελετηθούν. Ε, το θέμα αυτό μας απασχολεί διαρκώς και είναι ένα θέμα άμετα συνδεδεμένο με τα θέματα τα, τα τρέχοντα. ε, μιλήσατε για αυτούς που εκδίδουν τα CDS ε, και όχι μόνο ε, αυτούς που πληρώνουν. Πράγματι υπάρχει αυτή η διαφορά και το, το σημείο αυτό το οποίο επισημάνατε στο πλαίσιο της ε, ρύθμισης που κάνουμε που θα αποτελέσει τη βάση των συστάσεων που θα κάνουμε στο μέλλον είμαι έτοιμος να δουλέψω πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα με ένα απαραίτητο νομοθετικό μέσο. Ε, στον κύριο Χουντή. Ε, Βεβαίω ασκήσατε κριτική έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όταν βλέπετε το, τον αριθμό, το μέγεθος των κειμένων που βρίσκονται επιτάπητος, Πάντα μπορεί κανείς να πει ότι δεν ε, είναι αρκετά αυτά που κάνετε, δεν, ε, ε, δεν λειτουργείτε αρκετά γρήγορα. Μπορεί κανείς να ασκήσει αυτή την κριτική. Αλλά πράγματι υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος δεν μπορεί να συμπιεστεί. Είναι ο χρόνος των διαβουλεύσεων και πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις σε όλους τους τομείς, με όλους τους εμπλεκόμενους. Υπάρχει έργο τεχνικής φύσεως και νομικής φύσεως που πρέπει να ε, προηγηθεί. Σχετικά με το μη φύτα, ας πούμε, έχουμε ε, κείμενο 600 ε, σελίδων και κάθε λέξη, κάθε παύλα έχει το δικό της νόημα και τη βαρύτητα. Σχετικά με τους οίκους αξιολόγησης σας λέω σαφώς ότι αν κοιτάξετε το κείμενο που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την εξάρτηση των μεν από τους δε, διότι αυτό είναι το φοβερό. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν δηλαδή ε, αξιολογήσεις οι οποίες γίνονται σε όλους τους συσχετισμούς μεταξύ τραπεζών, εταιριών κλπ. Περισσότερος ανταγωνισμός. Θέλουμε να εξαλείψουμε όλους τους κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων και ε, βεβαίως ε, και το το θέμα της αξιολόγησης των ε, κρατών, αλλά επίσης και η υποχρεωτική έκδοση ε, των ε, συμπερασμάτων σχετικά με φορείς ή χώρες οι οποίες αξιολογούνται. Δεν είναι δυνατόν να, υπάρξουν, να υπάρχουν αξιολογήσεις χωρίς τις απαραίτητες εξηγήσεις. Σχετικά με τον ΟΤΕ, δεν θα επαναλάβω τα όσα είπα στην Ολομέλεια. Πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα το οποίο γνωρίζουμε καλά. Υπάρχει ε, ιδιωτικοποίηση που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα σεβαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα εφαρμόσει απολύτως τους κανόνες ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, Βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι μπορείτε να διατυπώσετε και ανησυχίες και διαφωνίες ως προς αυτό, αλλά δεν μπορώ να προσθέσω τίποτε παραπάνω. Ο κύριος Ανβέρ διατύπωσε νέες ιδέες με πολλή φαντασία, την οποία και εκτιμώ. Ε, είναι εφευρετικός, θα έλεγα. Και μου αρέσει αυτό. σχετικά με τα ΣΥΦΙΣ. Είμαι έτοιμος. να ασχοληθώ με αυτά, διότι σαφώς ομιλούμε δια οργανισμούς διεθνικούς και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης τι είναι ακριβώς το Financial Stability Board, υπό ποιες συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει, ποιο είναι το πεδίο δράσης κλπ. Και πρέπει να δούμε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί. Θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν, ας πούμε, τους κανόνες της Βασιλείας 2, καταρχήν. Ως προς την Βασιλεία 3 υπάρχουν τα οποία απαιτούν χρόνο και το θέμα της συμπληρωματικής κεφαλαιοποίησης που προτείνεται από κάποιους δεν είναι η μόνη απάντηση, δεν είναι η μόνη λύση. Υπάρχουν και άλλες α, λύσεις και μία εξ αυτών είναι τα σύφης. Είναι η εξωτερική εποπτεία, η εσωτερική εποπτεία, η διαχείριση της κρίσης κλπ. Και με μεγάλη χαρά θα ανοίξω τη συζήτηση αυτή στο πλαίσιο, το, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της συζήτησης του CRD4. Το είπα ήδη απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο με μεγάλη προσοχή θέλω να ξεχωρίσω το θέμα της διαχείρισης ε, κινδύνου, χωρίς καμία ιδεολογική προσέγγιση. Οι Βρετανοί αποφάσισαν να θέσουν το θέμα επιτάπητος με τις προτάσεις Βίκερς. Αυτά που προτείνει είναι προσαρμόσιμα στον τραπεζικό τομέα της ε, Παλαιάς Υπήρου. Και κοιτάζουμε τι κάνουν και οι Αμερικανοί. Και έχουμε έναν διάλογο και για τεχνικά θέματα και λειτουργικά με τον Τιμ Γκάιτνερ. αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως έγινε και με τον ε, Jacques Ντελαροζιέρ στο παρελθόν. Θα υπάρξει λοιπόν μια ομάδα εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό της δομής των τραπεζών και του διαχωρισμού της διαχείρισης κινδύνου και θα αναμένω τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας αυτής τους πρώτους μήνες. Διακόπτει ο μιλητής. Ε, θα πρότεινα στην ομάδα αυτή να υπάρχουν άνθρωποι από διάφορους τομείς και όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι σιγούνται την οικουμενική δομή τραπεζών, οι οποίοι θα, θα πούν ότι υπάρχει μία και μοναδική λύση. Κοιτάξτε, η Οικουμενική Τράπεζα, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ε, και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω ταμπού. Και θα το δείτε σε αυτό που κάνουμε στη Μυθήτα. Εγώ απαγόρευσα το trading από την πρώτη στιγμή. Ε, η ομάδα αυτή θα είναι αξιόπιστη και η εμπειρογνωμοσύνη της δεν θα αμφισβητείται, ούτως ώστε να έχουμε μια εντελώς, ε, ε, κάποια εντελώς αξιόπιστα συμπεράσματα βασισμένα στην εμπειρία τους. Και πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πεπειραμένοι σε αυτά τα θέματα και οι οποίοι πιστεύουν, οι οποίοι πιστεύουν στη ιδέα της Οικουμενικής Τράπεζας, οι οποίοι όμως θέλουν ασφαλώς να διαχωρίσουν το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου. Συγγνώμη, αν επιτρέπετε και άλλη μια ερώτηση στον Φιλίπ, θέλω και εγώ να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Το θέμα της μέγιστης εναρμόνισης δεν το θίγει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο προηγούμενος διοικητής, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας και ο κύριος Τελαρουζιέρ. Το να λέτε ότι το λένε μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία δεν, ε, δεν ισχύει. Και δεν είπα αυτό και δεν θέλω απάντηση τώρα, απλά θέλω απλά να αποκαταστήσω την αλήθεια. Γνωρίζω τις ε, βασικές ε, αρχές τις οποίες εσείς πρεσβεύετε και ο κύριος Τρισέ και ο κύριος Ντελαροζιέρ χρειάζονται ενθάρρυνση ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει εμπειρογνώμονες και αυτοί ασχολούνται και το κείμενο το οποίο παρουσίασα ε, τον Ιούνιο ε, αποφάνθηκαν ότι ήταν απολύτως σύμφωνο και συμβατό με τις αρχές της ε, Βασιλείας. Και επαναλαμβάνω ότι η ανάλυση που κάνουμε των δικών μας κειμένων για να τα βελτιώσουμε θα επιτρέπει την απαραίτητη ευελιξία ώστε κάποιες χώρες να προχωρήσουν πιο μακριά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαι δεσμευμένος να εκδώσω αυτό το single workbook ε, στο άμεσο μέλλον. Σχετικά τώρα με το shadow banking Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θέμα το, η επιβολή δηλαδή επιπρόσθετων ε, κανόνων στις τράπεζες. Το αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή όχι στο πλαίσιο του CRD4 δεν είναι απολύτως σαφές. Η Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα τέσσερις ε, ακόμα μιλητές ε, και παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί θα πρέπει να φύγει ο κύριος Επίτροπος και μετά τη τον διάλογο τον οποίο είχαμε τώρα, δεν νομίζω πως ε, χρειάζεται να περιορίζεται το Κοινοβούλιο για να ενσωματώσει ιδέες του στην τέταρτη οδηγία κεφαλιακής επάρκειας. Μάλιστα υπάρχουν πολλά πράγματα για μακροπροληπτικά εργαλεία και άλλα, τα οποία νομίζω θα θέλει να θίξει το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε αυτά που είπατε, δηλαδή την επιστροφή της πολιτικής μπροστά στη μοιοπία των αγορών. Έχουμε πολλά νομοθετήματα και γνωρίζουμε και τι μας είπατε τη Δευτέρα, τι είπατε τη Δευτέρα στον τύπο. Θα το αφήσω όμως αυτό στο Λεωνάρντο. Ως προς τη Βασιλεία 3 και το ΣΕΡΔΕ 4, εάν θέλουμε να κινηθούμε πιο γρήγορα από τις αγορές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όπως μας λένε οι υπεύθυνοι περί συγκυρίας, ότι θα φτάσουμε σε μια ε, γενικότερη επισφάλεια. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιδεινωθεί η φερεγγιότητα των τραπεζών, γιατί τότε θα αυξηθεί και το δημόσιο χρέος. Εάν λοιπόν οι τράπεζες θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι φερέγγες, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εκ νέου κεφαλαιοποίηση, στον αριθμητή αυτό. Όταν συζητούμε με τους τραπεζίτες μας λένε ότι στη γαλλική περίπτωση μπορεί να γίνει απορρόφηση της περίπτωσης Ελλάδας. Εάν όμως η Ιταλία δανείζεται με υψηλά επιτόκια, τότε θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα για αρκετές τράπεζες. Άρα υπάρχουν δύο λύσεις η πρώτοι να αποτανθούμε στις αγορές, αλλά όπως ξέρετε οι τράπεζες δεν μπορούν να εξεύρουν ιδίους πόρους και ίσως όπως το 2008 να ζητήσουμε την κρατική επιδότηση και εσείς είσαστε υπεύθυνο για να χορηγήσετε αδειοδότηση ή όχι. Μπορείτε να διατυπώσετε την ερώτησή σας, λέει η πρόεδρος. Ποια είναι η θέση σας προς το θέμα αυτό που αφορά την εφαρμοσιμότητα του ΣΕΡΔΕ 4 και της Βασιλείας 3. Ο Διόγκο. Ευχαριστώ. Σάρον, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ για αυτή την ε, πλαισίωση του θέματος που μας ε, εντυπωσιάζει. Πρόκειται για προτάσεις που έχουν υποβληθεί, μερικές έχουν ψηφιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για την δραστηριότητά σας σε αυτό τον τομέα. Μεταξύ των προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου που υποβλήθηκαν, ήθελα να σας συγχαρώ για την πρόταση ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήματα επί του θέματος. Το ένα θέμα έχει να κάνει με τη βαθμολόγηση των οίκων. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για την κατανομή της αγοράς και των αγορών μεταξύ των οίκων που έχουν ε, πολύ καλή φήμη και να δούμε πώς μπορεί να έχει αυτή η κατανομή. Ως προς την χρηματοδότηση των οίκων πιστοληπτικής ικανότητας, δεν ξέρω κατά πόσο νομίζετε ότι θα πρέπει να αλλάξει το πρότυπο χρηματοδότησης των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ικανότητας. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τον τομέα της εποπτείας, της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο η πρότασή σας θα ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της 12 η Σεπτεμβρίου, όπως μας τις εκθέσατε στην Ολομέλεια, ή κατά πόσο θα προβλέπονται άλλες δυνατότητες. Και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά τη στιγμή που διανύουμε μία περίοδο βαρύτατης της κρίσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα περιοριστώ στο θέμα των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα, κύριε Επίτροπε, μετά από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ρεαλιστής και να καταγράφει τις καταστάσεις όπως ορίζονται. Όμως δεν χωρεί αμφιβολία ότι έχουμε ένα νέο κανονισμό ο οποίος έχει αποδυναμωθεί κάπως ή έχει γίνει ανισόρροπο σε σχέση με την αρχική πρόταση. Θεωρείτε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις διατάξεις προς το καλύτερο και πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε ορισμένα θέματα δηλαδή ως προς την αναστολή βαθμολόγησης για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες. Και τι γίνεται ως προς τις συγχωνεύσεις ε, μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας των οίκων αξιολόγησης. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Εάν ναι, Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια κοινοβουλευτική εργασία που θα προβλέψει βασικές τροποποίησεις στις ε, διατάξεις αυτές. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα σαφές το πρότυπο που έχουμε κατά νου. Πιστεύετε ότι αν ίσχυε αυτός ο νέος κανονισμός, ας πούμε ότι είχε τεθεί σε ισχύ, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το σφάλμα των της Standard Poor's ως προς την αξιολόγηση της ε, Γαλλίας, ας το αποκαλέσουμε σφάλμα. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να δούμε θέματα όπως το δημόσιο χρέος, ε, την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για συγκρόμενα συμφέροντα, όπως είπε και ο συνάδελφος Φεγιό, και να δούμε και τι θα γίνει με έναν ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης. Επειδή είμαι εισηγητής, πρέπει να παρέμβω λίγο περισσότερο, Πρόεδρε. Συνήθως είμαι επιγραμματικός αλλά αυτή τη φορά πρέπει να μιλήσω λίγο περισσότερο. Σας υπενθυμίζω ότι η έκθεση Κλίντς αναφερόταν στον οίκο πιστοληπτικής ικανότητα σαν ένα ε, βασικό σημείο. Εδώ δεν γίνεται λόγος ούτε καν για εκπόνηση μελέτης αντικτύπου ε, στην οποία ε, επιδίδεται η ε, επιτροπή. Ε, δεν αφορούσε εσένα, Λιονάρντο. Είναι γενικό το θέμα. Ελίζα, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ. Συμφωνώ όταν λέτε ότι υπάρχει ο χρόνος των πολιτικών που είναι πιο μακροχρόνιος από τον χρόνο των αγορών. Νομίζω όμως ότι επειδή δεν είμαστε επαρκείς, δεν δείξαμε επάρκεια στις προτάσεις μας, δημιουργούμε ευκαιρίες έτσι ώστε να ε, είναι ηγέτες οι αγορές και όχι εμείς. Αναφέρομαι στο χρέος των κρατών και στα προβλήματα των τραπεζών. Νομίζω ότι οι μέτοχοι Διακόπτει ο μιλητής γιατί παρεμβαίνει κάποιος άλλος εκτός μικροφών. Ο Επίτροπος πρέπει να φύγει, αλλά αφήστε την Ελίζα να τελειώσει. Να συνεχίσω, λέει η Ελίζα. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Δηλαδή πρέπει να δούμε πρώτα το θέμα των κρατικών χρεών, του κρατικού χρέους ή των τραπεζών. Δεν πρέπει να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί ακόμα και οι χώρες υπό την Τρόικα μιλάνε για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές επιδεινούνται το χρέος που είναι ήδη πολύ βαρύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει επανακεφαλαιοποίηση αυτών των τραπεζών, δηλαδή των τραπεζών που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες υπό το πρόγραμμα της ε, Τρόικα. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση υπερβολικού χρέους. Για να μπορέσουν οι τράπεζες αυτές να αναλάβουν μέρο το, μέρος του χρέους θα πρέπει να γίνει επανακεφαλαιοποίηση η οποία να ακολουθεί πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Να γίνει μια επιτάχυνση δηλαδή της διαδικασίας γιατί μιλάμε για ε, τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν μέρος του κινδύνου. Άρα ε, μιλάμε για έναν φαύλο κύκλο ο οποίος υπονομεύει και τον ανταγωνισμό. Μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των τραπεζών σε κατάσταση κρίσης θα πρέπει να δούμε κατά πώς θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Ως προς το κρατικό χρέος τώρα όμως μιλάμε και για τη συμμετοχή της ΕΚΤ με την έκδοση ευρωομολόγων. Μέχρι όμως να γίνουν αυτά εκτιθέμεθα στα ratings στη βαθμολόγηση. Μπαίνουμε λοιπόν σε έναν ατέρμονο φαύλο κύκλο. Άρα η διαχείριση της τραπεζικής ε, κρίσης θα πρέπει να ε, εντάσσεται στο θέμα του δημόσιου χρέους. Βρισκόμαστε στο δημόσιο χρέος. Ε, άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού μέσα στα πλαίσια του, του φαύλου κύκλου. Έχετε το λόγο. Ναι, επειδή πιέζει ο χρόνος ε, δεν θα με Έχουμε όμως κάποια ανοιχτά ζητήματα. Εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Τα κρατικά ομόλογα σύμφωνα με την Βασιλεία 3 αξιολογούνται με κίνδυνο 0. Αποτελούν όμως ουσιαστικό πρόβλημα και θα μπορούσαμε ίσως ε, μέσω της ε, νομοθεσίας να αλλάξουμε αυτήν την αξιολόγηση 0 ε, με τριοπαθώς προς μια άλλη κατεύθυνση. Και θα πρέπει να συμφωνήσω πως έχετε επιδείξει όχι μόνο θάρρος αλλά και πραγματική εξοπιστία σε αυτό που και γι' αυτό έχει κερδίσει τον σεβασμό μα. Ε, τηλεγραφικά θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ όλου του παρεμβαίνοντε για τι ερωτήσει, αλλά και για την προτροπή και την ενθάρρυνση. Είπα και προηγουμένως στην κυρία Φόρνα, ε, πράγματι Θέλουμε να είμαστε απολύτως πιστοί στο πνεύμα και το γράμμα των συστάσεων της Βασιλείας ε, και ως προς το CRD4 και βεβαίως δεν έχει τελειώσει όλη η διαδικασία και ε, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και το τι ακριβώς συμβαίνει στις ευρωπαϊκές ε, οικονομίες. Ήδη έγινε αναφορά στο δημόσιο χρέος και εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό αυτό το έργο και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές επί του θέματος. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών που είπε ο Διέμ και η κυρία Φερέρα. Στην αρχή της παρέμβασής μου σας περιέγραψα το τι ακριβώς κάνουμε, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, για να έχετε μια σφαιρική εικόνα και το τι ε, αποφασίστηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 26-27 Οκτωβρίου. Εκεί καθορίστηκαν οι πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες και η πρώτη προτεραιότητα πέραν του ελληνικού ζητήματος, δηλαδή του αφόρητου ελληνικού κρέους ας πούμε, του, δημοσίου, του μεγάλου δημοσίου χρέους της Ελλάδος, υπήρχε και το θέμα των άλλων δημοσίων χρεών που απαιτούν την θέση σε ισχύ νέων μηχανισμών. Γι' αυτό λοιπόν από τη θέση στην οποία βρίσκομαι και τους συναδέλφους, τον Όλυ Ρέν, τον Ιωακή Μαλμούνια κλπ. Δουλεύουμε για να οθήσουμε παράλληλα τη θέση σε ισχύ όλων των αποφάσεων της 26ης. Όχι μόνο το θέμα της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η ανακεφαλαιοποίηση βεβαίως είναι ένα θέμα, αλλά θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση που διερχόμεθα, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και το θέμα του δημοσίου χρέους μέσω του Ταμείου Σταθερότητας. Και ο κύριος Γιάννοκ αναφέρθηκε σε αυτό, δηλαδή συντονισμό των χρηματοδοτήσεων μεσοπρόθεσμα. Το, ένα άλλο θέμα είναι το Ταμείο σταθερότητα για τα κράτη. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα ασφαλώς. Και δουλεύουμε σε όλα αυτά τα θέματα στη συνεργασία με τους Υπουργούς των Οικονομικών. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραματίζει το δικό της ρόλο από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της κρίσης και θα συνεχίσει να παίζει το ε, ρόλο της σύμφωνα με το καταστατικό της. Να πω επίσης ότι σε αυτή την ε, σφαιρική προσέγγιση το θέμα της ε, κεφαλαιοποίησης είναι ένα θέμα θεμελιώδες, αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση για την, ευρωστία των τραπεζ... την αποκατάσταση της ευρωστίας των τραπεζών. Υπάρχει και το θέμα της διακυβέρνησης, το θέμα της πρόληψης και επίλυσης της κρίσης. Όλα αυτά μαζί λοιπόν ως προς τον τραπεζικό τομέα. Ο κύριος φαγιό αναφέρθηκε στο θέμα των ε, εικοναξιολόγησης. Πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που συνέβη με τη Standard Poor's και τόσο οι γαλλικές αρχές όσο και οι χρηματοοικονομικές θέλουν να μάθουν ακριβώς το τι συνέβη. Ε, εγώ μάχομαι από αυτού πιστεύοντας βεβαίως ότι οι οίκοι αξιολόγηση είναι χρήσιμοι και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, χρήσιμο ρόλο. Και βέβαια υπήρξαν λάθη και σφάλματα και απαιτήθηκαν μεταρρυθμίσεις και έχουν γίνει αρκετές ε, τέτοιες ε, μεταρρυθμίσεις. Κάποιες αξιολογήσεις ε, κρατών κατέρευσαν δεν επαληθεύτηκαν δηλαδή και αυτό ακριβώς κλώνησε και την αξιοπιστία. Και εμείς θέλουμε αξιολογήσεις σαφείς, διαφανείς, εξηγήσιμες, που να στηρίζονται δηλαδή με την απαραίτητη με τις απαραίτητες εξηγήσεις. Μείωση της εξάρτησης, ενίσχυση του ανταγωνισμού, εξάλληψη των ε, συγκρούσεων συμφερόντων, μεγάλη προσοχή ως προς τα, το δημόσιο χρέος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί είναι και η αστική ευθύνη σε ούτως ώστε να επιβληθούν κυρώσεις όταν υπάρχουν όταν συμβαίνουν σφάλματα ή λάθη. Έτσι, έτσι ώστε οι αδυναμίες και τα προβλήματα που προέκυψαν στο παρελθόν να μην επαναληφθούν στο μέλλον με βάση τη νέα νομοθεσία. Η Κομισιόν με το έργο της αποδεικνύει ότι είναι ιδιαίτερα ε, προσεκτική αλλά και φιλόδοξη στην επιδίωξη των στόχων της. Κύριε Φαγιό, μιλήσατε ε, για το θέμα της χρηματοδότησης των οίκων αξιολόγησης. Δεν έχουμε ένα σύστημα ελεγχόμενης οικονομίας. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα μοντέλο πληρωμών. Όλα τα μοντέλα έχουν και τα θετικά και τα αρνητικά τους. αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια κάθε μοντέλου, κάθε προτύπου πληρωμής. Αυτό θεωρώ σημαντικό. Σχετικά με τον έλεγχο, συνεχίζουμε το έργο μας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε, δουλεύω υπό συνθήκες τις οποίες γνωρίζω καλά, δηλαδή αναπτύσσω μαζί με τους συνεργάτες μου τις προτάσεις με βάση την μέθοδο που ισχύει, δηλαδή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Και βλέπω διάφορα σχόλια στον τύπο. Γνωρίζω βέβαια πώς λειτουργεί, με επίτροπος πολλά χρόνια. Αλλά ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύεται εξαιτία διαρροής δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό, ενώ προβάλλεται ως οριστικό. Και αυτή είναι η δυσκολία μου. Εγώ θέτω ε, υπό διαβούλευση κείμενα και ακούω τις απόψεις συναδέλφων και ενδεχομένως με βάση αυτές τις απόψεις οι οποίες είναι απολύτως ε, ε, ορθές τα κείμενα αλλάζουν. Και όταν κάποιοι εξ αυτών εκφράζουν επιφυλάξεις ή ασκούν κριτική, ασφαλώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άλλο λοιπόν είναι το κείμενο το οποίο θα εμφανιστεί μετά από την διαβούλευση στο πλαίσιο της Κομισιόν και άλλο το, ένα κείμενο το οποίο διαρρέει από κάποια υπηρεσία. Και έχω πολλά τέτοια παραδείγματα και μπορώ να σας τα παρουσιάσω. Κείμενα δηλαδή της Κομισιόν τα οποία στην πορεία βελτιώθηκαν μέχρι να φτάσουν στη τελική τους μορφή. Ας πούμε σχετικά το, το κείμενο το σχετικό με τους ελέγχους και το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε σε επίπεδο G20. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια με περισσότερο ανταγωνισμό. Υπάρχουν ιδέες που εφαρμόζονται σε μία ή δύο χώρες Εν πάση περιπτώσει, τα, συζητούμε όλα αυτά. Θέλω απλώς να αποδραματοποιήσω την όλη συζήτηση και σας εξηγώ το πώς γίνεται η δουλειά σε επίπεδο συλλογικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι έδωσα επαρκείς απαντήσεις ε, ξεκάθαρες στο μέγιστο δυνατό βαθμό και περιμένω από εσά και την κριτική αλλά και την προτροπή και την ενθάρρυνση για να μπορέσω να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Επίτροπος θέλει να φύγει και μισή κύριοι συνάδελφοι, αλλά βεβαίως τελικά έλαβαμε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ.